και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Μυρίζει σε σάωνα. Και η θερμοκρασία επίσης θυμίζει σάωνα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Δεν μου αρέσει αυτή η μυρωδιά του ξύλου. Βέβαια, μου θυμίζει το Σαββατοκύριακο. Ο Κλοντ Μωράης βρίσκεται στη Ρουμανία στη συνεδρίαση της Europol, αν δεν κάνω λάθος, και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Κάτι που θα κάνω ευχαρίστω. Ξεκινάμε με την έγκριση μερίσιας διάταξης. Σημείο 1. Οι σοσιαλιστές και οι ΓΚΟΕ μου ζήτησαν να ψηφίσουμε δυνάμει του άρθρου 205, το σημείο 3,34 του ενημερωτικού σημειώματος για την απόφαση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα λάβουν οι συντονιστές στη συνεδρίασή τους. Αυτή θα είναι η πρώτη ψηφοφορία που θα έχουμε αύριο στις 12. Θα δώσω το λόγο όμως στην Πριγκίτε Ζίπελ για να μας εξηγήσει πού και πώς και γιατί. Όπως είπατε πολύ σωστά, θα ήθελα να αμφισβητήσω την απόφαση των συντονιστών να αποφασίσουν ε, μεταξύ τους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα σας εξηγήσω το γιατί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε μετά τη σχετική διάταξη της συνθήκης. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν λοιπόν να συστήσουν μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταπολεμήσουν την απάτη εις βάρος των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ξαφνικά, σαν παρόλο που το αποφάσισαν όλα τα κράτη-μέλη, τώρα μόνο 22 χώρε μέλη λαμβάνουν μέρο στη σύσταση αυτού του γραφείου τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ακόμη χειρότερο, ε, προσπαθούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε ότι όλη η διαδικασία έχει πολιτικοποιηθεί πλήρως. Και παρόλο που δεν αμφιβάλλω ότι οι υποψήφοι που έχουν υποβληθεί έχουν προσόντα και τα απαραίτητα εφόδια, ε, με ενοχλεί αυτή η πολιτικοποίηση της διαδικασίας. Ένα από τα τελικά σημεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα τελευταία μας ε, θέματα, είναι να αποκαταστήσουμε μία διαφάνεια, όχι μόνο οργανώνοντας δημόσια ακρόαση, αλλά και ψηφίζοντας το συγκεκριμένο υποψήφιο, ένα κατάλογο υποψηφίων, στην ολομέλεια τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και όχι και κλεισμένο το θηρό να γίνει ψηφοφορία μόνο μεταξύ των συντονιστών. Αμφισβητώ λοιπόν και ε, ενίσταμε για αυτή την απόφαση των συντονιστών να αποφασίσουν μεταξύ του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητώ να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αύριο, μάλιστα. Οπότε αύριο θα ψηφίσουμε αυτό το αίτημα στις 12. Ε, και γιατί ακριβώς εδώ και τώρα να εξηγήσουμε. Παρόλο που είμαι ε, ε, αναπληρώτρια εδώ ε, πρόεδρος, ε, η ένσταση για μια διαδικασία απαιτεί και προφορική εξήγηση, όχι μόνο γραπτή. Γι' αυτό σα έδωσα το λόγο και σα ευχαριστώ που μα ενημερώσατε. Περάμε τώρα στο σημείο, να σα πω ότι το σημείο 18, μάλλον το σημείο 17 τη ημερήσια διάταξη, Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι «Ε, χρειάζονται βίζα για να περάσουν τα εξωτερικά σύνορα κτλ. κτλ. Αναβάλλεται. Το σημείο 17 λοιπόν αναβάλλεται. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Τώρα, γλωσσικό καθεστώς. Θα έχουμε διερμηνία από και προς όλες τις γλώσσες με εξαίρεση τα μαλτέζικα, κροατικά και ιρλανδικά αγωγελικά. Ε, προχωρούμε στην έγκριση των συστάσεων των συντονιστών δυνάμει του άρθρο 205. Ε, το ενημερωτικό σημείο με τη συνεδρίαση της 19 Φεβρουαρίου του 2019 υπάρχει στα έγγραφα της συνεδρίασης και όπως είπαμε στο σημείο 1, το ενημερωτικό σημείωμα των συντονιστών υποβάλλεται στην Επιτροπή για έγκριση με εξαίρεση το σημείο 3, σημείο 4, για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Είχαμε και διορισμό εισηγητών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λίβε ε, αναλαμβάνει ε, το σχέδιο ψηφίσματος για την ανακοίνωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για μια Ευρώπη που προστατεύει και την προστασία να επεκταθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Συγγελίας στο διασυνοριακό τρομοκρατικό έγκλημα. Ελπίζω να εγκρίνετε τι συστάσει των συντονιστών με εξαίρεση το 3-4, όπω είπαμε, για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Και επαναλαμβάνω ότι η ψηφοφορία για το 3-4 θα γίνει αύριο στι 12. Οπότε μην ξεχάσετε, παρακαλώ, τι κάρτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε εγκρίνει και τα πρακτικά τη της 10 Δεκεμβρίου, της 4 η Ιουνίου, 26 Φεβρουαρίου, όχι γιατί είναι αυτή η σημερινή και αυριανή. Α, του 2018, 26 27 Φεβρουαρίου 2018 και 11 και 12 Οκτωβρίου 2017, πολύ παλιά πρακτικά. Αλλά εγκρίνονται και αυτά. Και περνάμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημέρης διάταξης, το σημείο 4, η θέσπιση του προγράμματος για τα δικαιώματα και τις αξίες. Μετά την έγκριση της εντολής ε, τον Ιανουάριο του 2019 στην Ολομέλεια έγιναν τρεις τρίμερες διάλογοι, 22 Ιανουαρίου, 5 Φεβρουαρίου και 20 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μποντήλ Βαλέρο που θα λάβει και το λόγο για να μας παρουσιάσει για λίγα λεπτά το πρόγραμμα αυτό και να μας κατατοπίσει. Παρακαλώ κυρία Βαλέρο. Mm. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους, ε, την συνεισηγήτριά μου, την κυρία Σύρπα είναι από την Επιτροπή Γυναικών και την κυρία Σιλβίκη Γιώμα, την Επιτροπή Πολιτισμού. Είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία με τις δύο συνεισηγήτριες και να ευχαριστήσω φυσικά και τους σκιώδεις συγητές, τη γραμματεία, τους συμβούλους και τους βοηθούς μας, γιατί ήταν πραγματικά πολύ αξιέπαινη και η δική τους προσπάθεια. Όπως είπατε, είχαμε ήδη τρεις τριμέρεις διαλόγους για το πρόγραμμα αυτό. Το Μάιο λάβαμε πέρυσι την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υιοθετήσαμε εμείς το σχέδιο εκθεσής μας το Δεκέμβριο του 2018 και το ίδιο έκανε και το Συμβούλιο και κατόπιν ξεκίνησαν οι τριμερείς διάλογοι τον Ιανουάριο έγινε ο πρώτος. Όπως είπατε, μέχρι στιγμής διεξήγησαν τρεις τριμερείς διάλογοι. Ο πρώτος για να έχουμε μια βολιδοσκόπηση των μερών για τις απόψεις τους. Το Συμβούλιο όμως ακόμη δεν έχει λάβει εντόλη για τα πιο σημαντικά θέματα. Και εμείς ζητήσαμε ένα νέο σκέλος για τις αξίες στο νέο πρόγραμμα γιατί το πρόγραμμα αυτό συγκερνά τα προηγούμενα ουσιαστικά και εμεί θέλαμε ένα νέο για τις αξίες. Επίσης, προτείναμε το μηχανισμό στήριξη των αξιών. Στον τελευταίο τριμερή διάλογο έγινε συζήτηση με το Συμβούλιο και με πολύ χαρά μπορώ να σας ενημερώσω ότι το τουλάχιστον το σκέλος των ενωσιακών αξιών είναι, προχωρά καλά. Φαίνεται δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα δούμε τώρα πώς θα το παρουσιάσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο στο διατακτικό. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη. Πάντως είναι θετικό ότι δέχτηκαν αυτό το νέο σκέλος για, την, για τις ενωσιακές αξίες. Τώρα το θέμα είναι πιο δύσκολο σε ό,τι αφορά το μηχανισμό στήριξης των αξιών. Πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε και ο μηχανισμός στήριξης των αξιών να συμπεριληφθεί στο νομικό κείμενο. Όπως είπα, το Συμβούλιο έχει λάβει πια την εντολή για να εξετάσει το νέο σκέλος, το νέο τμήμα για τις αξίες, αλλά για το υπόλοιπο τμήμα θα πρέπει να περιμένουμε. Επίσης, έχουμε διεκπαιρεώσει τη συζήτηση για πολλά άρθρα, μερικά και οριζόντιου χαρακτήρα, όπως το άρθρο 1, το πεδίο εφαρμογή, το 4, η συμμετοχή των πολιτών και ε, το θέμα της συμμετοχής γενικώ, ε, που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτισμού, άρθρο 9, για τη θέσπιση της ομάδας ε, πολιτικού διαλόγου και άλλες οριζόντιες διατάξεις. Ο νέο επόμενο τριμερής διάλογος θα γίνει σε 6 Μαρτίου, θα είναι ο τέταρτος και ελπίζω εκεί να διεκπαιρεώσουμε και τα τελευταία εκκρεμή σημεία της συζήτηση. Ευελπιστώ τουλάχιστον. Βέβαια κάποια καθόδη σημεία έχουν μείνει εκκρεμή, όπως είναι ο μηχανισμός για τη στήριξη των αξιών. Πάντως η συζήτηση γίνεται σε ευχάριστο κλίμα και πολύ επικοδομητικό πνεύμα γιατί και τα τρία θεσμικά όργανα θέλουν να εγκρίνουν και το μηχανισμό στήριξη για το νέο πρόγραμμα αλλά και το σύνολο του προγράμματος. Οπότε είμαι αισιόδοξη, θα βρούμε λύση. Ευχαριστώ.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 Λοιπόν, συμμετοχή των πολιτών, η Ευρώπη των πολιτών πραγματικά έχει μεγάλη σημασία, είναι κεφαλαίου σημασία, διότι είναι ένα πρόγραμμα πασίγνωστο, ε, το εκτιμούν πολύ, είναι κοντά στους πολίτες και εκφράζει την ε, πολίτη, την Ευρώπη, την καθημερινότητα. Λοιπόν, πρέπει και δίνει σάρκα και οστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θέλουμε να το προωθήσουμε το θέμα και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα διεξάγοντας τις συζητήσεις με ένα πνεύμα προσοχής και α, ε, σύνεσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αντικαθιστώ της και ο για το θέμα τον Μάικλ Μπόνιο που δεν μπορεί να παραστεί. Ο Μάικλ θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια την Ποντίλ Βαλέρο για τις προσπάθειές της. Σημαντικότατο θέμα, άριστη συνεργασία και συνεδρίαση των σκιωδών και στις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου. Οι συνάδελφοι όλων των μεγάλων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου είναι συντονισμένοι στις διαπραγματεύσεις και έτσι στην κοινωνία των πολιτών των 100 μελών στέλνουμε ισχυρό μήνυμα που θέλουμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες και θέλουμε να στηρίξουμε μια υγιή ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία προχωρήσαμε την περασμένη εβδομάδα με το Συμβούλιο μπορεί να διαπραγματευτεί το νέο σκέλο που αφορά τι οργανώσει κοινωνία των πολιτών που κινούνται σε αυτό το τομέα και θέλουμε να προωθήσουμε τι ευρωπαϊκέ αξίε όλα τα επίπεδα, αλλά όλο ιδιαίτερο στο τοπικό επίπεδο. Αυτό ήταν το βασικό θέμα το οποίο θέλαμε να πετύχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η σκιώδη εισηγητή είναι πολύ ικανοποιημένο που τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και να επεξεργαστούμε το τελικό κείμενο που αφορά αυτό το σκέλο. Η Σοφή Ιντφελτ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για όλη τη δουλειά που έκανε και κάνει. Ε, υποστηρίζουμε ολόθερμα ε, το ότι τονίζεται αυτό το νέο σκέλος. Έχω κάποιο σχόλιο σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των τριμερών διαλόγων μέχρι τώρα και το μηχανισμό στήριξης των αξιών που είναι ένας μηχανισμός υποστήριξης για τις ΜΚΟ σε χώρες όπου υπάρχουν πολλές πιέσεις εναντίον αυτών των φορέων. Δεν θέλω να κατονομάσω χώρες όπου αυτό ισχύει, που δέχονται πιέσει ΜΚΟ. Ε, να αναφερθώ καταρχάς στη διεξαγωγή των τριμερών διαλόγων. Εξεπλάγει από τη μεγάλη παρουσία και την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι θεωρώ ότι υπάρχουν δύο νομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που το εκπροσωπεί η Προεδρία του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μόνο δυνατότητα να αποσύρει μια πρόταση. Αλλά είναι αστείο να βλέπει κανείς πώς κυριαρχεί στη συνομιλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεσπόζει και επί της Προεδρίας και πιέζει το δικό της πρόγραμμα. Αυτός δεν είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά, όσον αφορά τον μηχανισμό υποστήριξη των αξιών, είναι σαφέστατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία όρεξη για κάτι τέτοιο. Ενώ το Συμβούλιο το ίδιο δεν είναι τόσο αμετακίνητο. Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να έχει υπόψη της ότι διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο, ε, όχι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι έχουμε υθετήσει μια θέση και ότι ο μηχανισμός υποστήριξης των αξιών που παρεπιπτόντος ήταν κάτι που απέρευσε από τις προτάσεις του κυρίου Μπόνι του ε, του ΕΛΚ ότι είναι κάτι που επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμη πιο ξεσημείωτο αν θεωρήσει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη της δημοκρατίας ε, και των αξιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε μηχανισμό κατεπίγουσης ανάγκης και δεν έχουμε τελικά τέτοιο μηχανισμό εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι παράδοξο, θα έλεγα. Θα ήθελα λοιπόν ο, η συγγήτρια να επιμείνει πολύ από αυτού. Βέβαια, κατά διάρκεια των πραγματεύσεων πάντα κανεί μπορεί να βρει δημιουργικέ λύσει. Δεν θα πρέπει να είναι αυτολεξή το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα περάσει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμη σημασία και πραγματικά πιστεύω ότι αν το τελικό κείμενο δεν εμπεριέχει αυτέ, αυτό το μηχανισμό υποστήριξη των αξιών, θα είναι πολύ πιο αδύναμο από αυτό που αρχικά ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Σεσίλ Κέγκε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τζούντιθ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Μποντίλ. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να πω ότι η επεξεργασία των τροπολογιών και εξέταση των επιχειρημάτων που υπευλήθησαν στις πολιτικές ομάδες ε, έγινε με πολύ σωστό τρόπο, ελήφθησαν όλες οι απόψεις υπόψη είχαμε μια ιδιαιτερότητα και θέλαμε να επιμείνουμε επί της αναγνωρίσεως άλλων μορφών διακρίσεως. Κάτι που αναγνωρίστηκε και εντό του κειμένου. Ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, καταπολέμηση της βίας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου και ήθελα να πω ότι όλες οι τροπολογίες που υπευλήθησαν εγκρίθηκαν. Χαίρομαι για αυτή τη νέα συνάντηση που ανέφερε, για το νέο τμήμα μάλλον που ανέφερε η συγγήτρια για τις αξίες. Λυπάμαι μόνο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όσον αφορά το μηχανισμό υποστήριξης των αξιών, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στην εισηγήτρια, είμαι σίγουρη ότι όσο μας αφορά και σαν πολιτική ομάδα, είμαι σίγουρη ότι η εισηγήτρια θα βρει ευνοϊκό έδαφος για να περάσουμε αυτές τις απόψεις. Την εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τη δουλειά που έκανε. Αυτή η δουλειά για μας είναι σημαντικότατη, διότι για πρώτη φορά προβλέπουμε και μηχανισμό χρηματοδοτήσεως που συνδέεται με τις αξίες. Αξίες που αναφέρονται εδώ στο κειμένο και πιστεύω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό κείμενο πολιτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αραγέ στη θέση του και αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλά σημεία. Ό,τι θέλαμε να προωθήσουμε και έπρεπε να περάσουμε έτυχε τη ίση υποστήριξη, είχε συντονιστεί το Κοινοβούλιο. Και χάρη βέβαια στη δουλειά τη Μποντίλ, τη συνεργασία με τι πολιτικέ μα ομάδε. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο. Θα επιτρέψω να λάβετε το λόγο. Θα σας παρακαλούσα όμως λάβετε υπόψη αυτό που είπε και η Σοφή Ιντεφέλτ. Και αν σαν προσωρινή πρόεδρος να πω ότι δεν υπονοείται ότι αυτόματα θα τοποθετείτε το, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ενημερώνετε τα μέλη του Κοινοβουλίου σε πραγματεύσεις. Είναι πολυτέλεια που μπορείτε δημόσια να ακούσετε την ενημέρωση που κάνει η συγγήτρια ε, στους άλλους συναδέλφους. Μαρία Τόμασέτη, έχοντας αυτό υπόψη, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω ότι δεν ζητήσαμε το λόγο. Από εσά εξαρτάται. Ευχαριστώ πολύ. Θα σταματήσουμε εκεί. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, αύξηση Μποντήλ, α, συγγνώμη, έχεις το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Να απαντήσω στη Σοφή. Όπως το είπες, έτσι είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει αυτό να το προωθήσει. Και δίσταζε και το Συμβούλιο. Αλλά γνωρίζω ότι στο Συμβούλιο, στη συζητήση του Συμβουλίου, υπήρξε μεγάλη αντίσταση. Όπως είπες, δεν θα είναι η ίδια κατάσταση, δεν θα έχουμε το ακριβές κείμενο που ζητήσαμε. Ζήτησα όμως κάποιες δημιουργικές λύσεις. να δούμε πώς να βρούμε μια διεξοδό για να έχουμε αυτό το μηχανισμό υποστήριξη των αξιών. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν πιστεύω όμως ότι θα έχουμε το ίδιο κείμενο που είχαμε αυτό που προτείναμε. Δεν θα είναι το ίδιο ακριβώς κείμενο αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε φτάσει, έχουν καταλήξει στο τελικό κείμενο ακόμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Συγγνώμη που σας ξέχασα. Περνάμε τώρα στο σημείο 5, την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητα των Ευρωπαίων πολιτών και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους κατά, κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης. Ο κύριος ε, Πρέ είναι ο εισηγητής και έχει και το λόγο για λίγα λεπτά για να μας παρουσιάσει αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν ε, πρόσφατα στις 19 Φεβρουαρίου ε, με ακρίβεια ε, για μια προσωρινή συμφωνία επί του θέματος ε, που αναφέρατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους κοιόδης κυρίως των πολιτικών ομάδων για τις πολύ ευρυθείς ε, σοβαρές μεστές συζητήσεις που είχαμε παρά τις κάποιες διαφωνίες και τις πολύ θερμές εγκάρδιες συζητήσεις. Και ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής μας, τους συμβούλους πολιτικής των διαφόρων ομάδων και τους βοηθούς μας. Ποιο είναι ο στόχο αυτή τη πρόταση, καταρχήν, κυρία Πρόεδρε. Στόχο τη πρόταση είναι να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των μελών τη οικογένειά του, ενισχύοντα τα στοιχεία τη ασφάλεια των δελτίων ταυτότητα και των ε, εγγράφων διαμονή. Πρωταρχικό μα στόχο είναι να διευκολύνουμε την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Θα ήθελα καταρχήν να σας διευκρινίσω τι δεν είναι η πρόταση αυτή. Δεν δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό δελτίο ταυτότητας παράλληλο με τα εθνικά δελτία ταυτότητας. Δεν αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη που δεν εκδίδουν δελτία ταυτότητας να το κάνουν από εδώ και πέρα. Ούτε δημιουργούμε μια τράπεζα δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, ο προτινόμενος κανονισμός επουδενεί δεν αποτελεί νομική βάση για τη ε, δημιουργία βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά να τα διευκρινίσω. Τι δεν είναι η πρόταση, τι δεν είναι ο κανονισμός. Αυτό που επιδιώξαμε πέραν της αρχικής πρόβλεψης της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητα και το επανάγνωστο των δελτίων ταυτότητας, γιατί έτσι θα διευκολύνουμε όντως την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Οπότε, αν συμφωνήσετε για αυτή την προσωρινή συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, θα έχουμε ένα πια ενίο πρότυπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα δελτία ταυτότητα. και θα, θα αναφέρονται τα ίδια σημεία με συγκεκριμένη σειρά επίσης για να είναι πιο ευανάγνωστα αυτά τα δελτία ταυτότητας. Επίσης όπως ε, ισχύει και για τις άδειε οδήγηση και για τα διαβατήρια, θα έχουμε και ένα ευρωπαϊκό σύμβολο. Σε ό,τι αφορά την αναφορά του φύλου, καταφέραμε να είναι προαιρετική αναφορά του φύλου στα δελτία ταυτότητας. Επίσης, ε, θα αναφέρεται η λέξη gender και θα υπάρχουν τρία, ε, τρεις το X, το F και το M, για τον προσδιορισμό του φύλου, του gender. Επίσης, ε, θα πρέπει όλα τα δελτία ταυτότητα να αναγνωρίζονται υποχρεωτικά ως έγκυρα έγγραφα σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις χώρες. Επίσης, καταφέραμε να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας των δεδομένων και να ενισχύσουμε την ευθύνη των κρατών μελών για την τήρησή τους. Υπάρχουν σαφείς μνήες στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων, το GDPR. Επίσης υπάρχει σαφής περιορισμός της πρόσβασης στα βιομετρικά δεδομένα μόνο στο προσωπικό, στο διαπιστευμένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών και μόνο προκειμένου να εξακριβώσουν τη γνησιότητα του εγγράφου και την ταυτότητα του δικαιούχου του. Επίσης, προβλέπεται σαφέστατα ότι τα βιομετρικά στοιχεία δεν ε, θα κρατούνται παρά μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά του τσιπ και με βάση περιπτώσει στη συνέχεια θα πρέπει να καταστρέφονται. Εκτός και αν λόγω της εθνικής νομοθεσίας και πέραν των δικών μας αρμοδιοτήτων κάποια κράτη-μέλη κρίνουν απαραίτητη την ε, ε, κατοχή αυτή, την παρακράτηση αυτή των δεδομένων προκειμένου να συστήσουν μια τράπεζα δεδομένων. Αλλά αυτό είναι δική του αρμοδιότητα, δεν μπορούμε να του εμποδίσουμε. Επίση, προβλέπουμε σαφέστατα ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ακαιρεότητα, την αυθεντικότητα, την γνησιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν ιδιωτικέ εταιρείε για την έκδοση αυτών των δελτίων ταυτότητα. Οπότε εξακολουθούν να είναι πλήρω αρμόδια και υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων. Το πιο λεπτό και ευαίσθητο σημείο των διαπραγματεύσεων, κυρία Πρόεδρε, ήταν το κατά πόσο τα δακτυλικά αυτά αποτεπώματα θα είναι υποχρεωτικό να λαμβάνονται σε όλα τα κράτη-μέλη που χορηγούν δελτία ταυτότητα. Ή θα αφήναμε τη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν λοιπόν κατά το δοκούν αν θα τα συμπεριλάβουν ή όχι. Δεν σα κρύβω ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε με στένος την προαιρετική αυτή δυνατότητα. Βέβαια, δεν καταφέραμε να ε, κυριαρχήσει η δική μας άποψη για λόγους ασφάλειας και ε, για το να είναι πιο ευανάγνωστα τα δελτία ταυτότητας. Γιατί σε περίπτωση που ήταν προαιρετική η συμπερίληψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν θα είχαμε το, τις ίδιες πληροφορίες σε όλα τα δελτία ταυτότητας. Κάτι που δημιούργησε πρόβλημα και ως προς την αναγνωσιμότητα και την ε, αναγνωρισιμότητα των δελτίων ταυτότητας. Γι' αυτό τελικά συμφωνήσαμε παρά τι επιφυλάξει κάποιων αντιπροσωπιών. Συμφωνήσαμε λοιπόν να έχουμε ακριβώς το ίδιο που ισχύει για τα διαβατήρια. Γιατί όπως ξέρετε τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι υποχρεωτικά στα διαβατήρια που χορηγούνται, εκδίδονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, καταφέραμε να συμφωνήσουμε και τη διάρκεια της ε, εφαρμογής αυτού του μηχανισμού και τη σταδιακή αντικατάστασης των παλιών δελτίων από τις καινούργιες ταυτότητες που θα πληρούν τους νέους κανόνες που σας προανέφερα. Θεωρώ ότι κερδίσαμε όσα μπορούσαμε, ό,τι μπορούσαμε το καταφέραμε και θα ήθελα να συστήσω στην Επιτροπή μας να εγκρίνει τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος κυρία Σαρτζεντίνη. Κάρλος Κουέλιο, σκιώδης ηγητής του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Ζεράρ Πχε για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε. Ήταν πραγματικά θριαβευτική νίκη για την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα ήταν σημαντικό να ενισχύσουμε την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονή και ταυτόχρονα θα επιδιώξαμε μια σύγκληση μεταξύ των Ευρωπαίων και τη διευκόλυνση όσων διακινούνται στο χώρο Σέγγεν. Επίσης θέλησαμε να διατρανώσουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και γι' αυτό έχουμε τα, κάποια οπτικά στοιχεία όπως τη σημαία που συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Στην πατρίδα μου την Πορτογαλία Εκατοντάδες χιλιάδες ε, πολίτες μετακινούνται στο χώρο Σέγγεν και είναι σημαντικό να γίνει σεβαστή η εθνική δελτία ταυτότητας, το εθνικό δελτίο ταυτότητας ε, που έχει μια πολύ σημαντική υπεραξία. Επίσης, ε, είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα δεκτυλικά αποτυπώματα και άλλα στοιχεία ασφάλειας. Γιατί έτσι όχι μόνο θα βελτιώσουμε τη, τα δελτία ταυτότητας, αλλά θα προστατεύσουμε καλύτερα και τα παιδιά μας. Όπως είπε και ο κύριος Ζεράρ Ντεπρέ, αυτό δεν θα επιβαρύνει ε, πλέον τους πολίτες. Δεν υπάρχει πρόσθετο κόστος, ούτε και επιπλοκές. Γιατί όταν θα χρειαστεί να ανανεώσουν την παλιά τους ταυτότητα, θα λάβουν την καινούρια. Δεν χρειάζεται να σπεύσουν να το κάνουν νωρίτερα. Επίσης, κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν κατά της συμπερίληψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Απλώς ήμασταν κατά της υποχρεωτικής ε, συγκέντρωσης των δακτυλικών δακτυλικών αποτυπωμάτων. Δεν θέλαμε να τα απαγορεύσουμε, αλλά να αφήσουμε τη διακριτική ευκαιρία στα κράτη-μέλη για τη συλλογή αυτών των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όλο παραδόξω, ε, τα κράτη-μέλη προτίμησαν οι Βρυξέλλε να λάβουν αυτή την απόφαση. Η συμφωνία αυτή είναι ισορροπημένη, έχει θεμελιώδη αξία για την ενίσχυση ευρωπαϊκή ηθαγένεια και διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και μάλιστα με ασφάλεια. Συγχαρητήρια, κύριε Ζεράρντε Πρέ. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Κάουφμαν, σκιώδη εισηγήτρια συγγνώμη, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω Λίαν Εγκαρδίος, τον εισηγητή μας, κύριο Ντεπρέ. Αληθεύει αυτό που είπε, ότι η συνεργασία πήγε πολύ καλά, ήταν πολύ εντατική μπορέσαμε να συζητήσουμε με αντικειμενικό τρόπο και με συντροφικό τρόπο πολλά θέματα. Βεβαίως πολιτικά ξεκινούμε από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά το έργο του, δηλαδή να υποστηρίξει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το επετέλεσε πολύ καλά. Και στις διαπραγματεύσεις του Συμβούλιο επίσης και τον ευχαριστώ ιδιαίτερω. Είπε ο Ζεράρντε Πρέ ότι επιτύχαμε πολλά. Δεν θα τα επαναλάβω αυτά που εξήγησε, αληθεύει όμως αυτό που είπε. Αν μου επιτρέπετε ωστόσο, επανέρχομαι σε αυτό το ακαθόδες θέμα που έτσι το περιέγραψε και ο ίδιος. Για μένα είναι μια θλιβερή νότα το γεγονός ότι περιλαμβάνουμε στο κείμενο την υποχρεωτική συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων στι χώρε μέλη. Ω Επιτροπή αντιταχθήκαμε ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή και για τη δική μου πολιτική ομάδα ήταν σημαντικό το θέμα αυτό. Σε όλε τι συζητήσει που διεξαγάγαμε από πλευρά Συμβουλίου, κατά τη γνώμη μου, κανένα απολύτω πιστικό επιχείρημα δεν μπόρεσε να προβάλλει το Συμβούλιο γιατί άραγε είναι αναγκαία η υποχρεωτική συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων πέραν των άλλων βιομετρικών δεδομένων. Εγώ θεωρώ ότι το μέτρο αυτό δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι αναλογικό και δεν υπάρχουν άλλωστε ούτε αριθμοί που να δείχνουν ότι δήθεν οι ταυτότητες που φέρνουν δακτυλικά αποτυπώματα είναι πολύ πιο ανθεκτικές απέναντι σε προσπάθειες πλαστογραφησής τους. Είπε και ο κύριος Κέλιο ότι δύο τρίτα των χωρών μελών δεν γνωρίζουν την υποχρεωτική συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και άλλωστε, είναι προφανές ότι οι χώρες μέλη θα θέλουν να ρυθμιστεί αυτό από τις Βρυξέλλες. Για την Γερμανία πάντως το θέμα δεν συζητείται. Δηλαδή δεν ε, το συζητεί το κοινό. Εθελοντικά μπορούμε να δώσουμε δακτυλικά αποτυπώματα εάν θέλουμε να ζητήσουμε νέα ταυτότητα. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Πάντως, ως πολιτική ομάδα δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με την ε, ε, τελική θέση που προέκυψε από, τις, ε, από τους τριμερείς διαλόγους. Ο σκιώδης εισηγητής των Πρασίνων, ή μάλλον η σκιώδης εισηγητρία, η κυρία Ζολή, είναι απούσα Πάντω έχει στείλει, μας έχει στείλει ένα μήνυμα στο οποίο ευχαριστεί τον κύριο Ντεπρέ και ζητεί να πούμε ότι η πράσινη δεν είναι ικανοποιημένοι με την έκβαση σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και το EDPS και ο Οργανισμός των Θεμελιών Δικαιωμάτων είναι επίσης αντίθετη. Η δε μελέτη δικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τα αποτυπώματα ως πρώτη επιλογή. Μόνο 10 χώρες μέλη το προβλέπουν αυτό στην νομοθεσία τους. Και δεν είναι εκπληκτικό που αυτή ήταν και η έκβαση των συζητήσεων με το Συμβούλιο, εφόσον μόνο 10 από τις 28 χώρες μέλη έχουν την υποχρέωση αυτή στην νομοθεσία τους. Κύριε Ντεπρέ, θέλετε να επανέλθετε έχοντας ακούσει τους ε, σκιώδεις συνεισηγητές σας ή θέλετε να ολοκληρώσουμε. Αν θέλετε να επανέλθετε μπορώ να σας δώσω ένα λεπτό ακόμη και μετά θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ασφαλώς αυτό ήταν το δύσκολο θέμα όπως είπε η κυρία Κάουφμαν. Ακούγοντας και την ανάγνωση της επιστολής της κυρία Ζολή υπενθυμίζω για ποιο λόγο επέμεινα στη διάρκεια τριών τριμερών διαλόγων. Όμως, το Συμβούλιο δεν δέχτηκε να μετακινηθεί από την θέση του και είπα εγώ τότε ότι το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί. Και τοποθετήθηκε το Κοινοβούλιο. Μπορεί να ακουστούν επιχειρήματα και προ τη μια και προ την άλλη κατεύθυνση. Όμω, ας μου εξηγήσει κάποιο αντικειμενικά για ποιο λόγο για τον Ευρωπαίο πολίτη θα δεχόμασταν δήθεν να περιλαμβάνονται τα δεκτικά του αποτυπώματα στο διαβατήριο, όχι όμω την ταυτότητα, στο δελτίο ταυτότητα. Και αυτό έχει γίνει δεκτό. Σαρτζεντίνη, σα ευχαριστώ. Εάν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι συμφωνήσουν στι 27 Φεβρουαρίου με την έκβαση των ε, τριμερών διαλόγων, η Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών θα ψηφίσει τότε στι 11 Τρίτου και πιθανότατα το θέμα αυτό θα έρθει στην Ολομέλεια στην δεύτερη περίοδο συνόδου του Απριλίου. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά και προχωρώ στο υπαριθμό 6 της ημερησίας διατάξεως. Δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σρόντερ, εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Εκπαίδευσης για τις αρχές επιβολής του νόμου βρίσκεται κοντά μας σήμερα για να εξηγήσει τα πορίσματα της πρώτης αξιολόγησης που έχει κάνει ο οργανισμός του για την ΣΕΠΟ και σας παρακαλώ να καθίσετε κύριε Σρόιντερ πριν να σας δώσω το λόγο. Υπενθυμίζω ότι ε, μόλις σας διανύμαμε ένα ε, φυλάδιο. Έχει το λόγο κύριε Σρόιντερ Μια στιγμή όμως Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Βεβαίω δεν είστε υποχρεωμένο να τα εξαντλήσετε τα 10 αυτά λεπτά, αν δεν τα χρειάζεστε. Αρχίστε όμω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μείνω στα 10 λεπτά, αφού σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι ενώπιόν σας και ευχαρίστω σα παρουσιάζω ορισμένα από τα απορίσματα τη έρευνα, αλλά και το τι θα κάνουμε για το 2019. Να ακολουθήσει η επόμενη διαφάνεια. τι πετύχαμε το 2018, τι έχει κάνει η ΣΕΠΟΛ που σχετίζεται άμεσα με τη συνεργασία με τις ε, αρχές επιβολής του νόμου. Έχω δύο παραδείγματα. Μιλούμε για την άμεση για τα άμεσα αποτελέσματα και για joint investigation teams, δηλαδή με αξιωματούχους που συμμετέχουν σε κοινέ ε, ομάδες ερευνών και σε συνεργασία με χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και με Ευρωπαίου Αξιωματούχου, που διαπιστώσαμε στην εκπαίδευση ότι αντιμετωπίζουμε τι ίδιε εγκληματικέ ομάδε. και προχώρησαν μετά σε έρευνε μαζί οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτέντε. και ένα άλλο παράδειγμα είναι το βίντεο training για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό των θυμάτων και την άμεση διάσωσή τους. Σας δείχνω με τον τρόπο αυτό πώς ο οργανισμός μας υποστηρίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και ποιες επιχειρησιακές επιτυχίες έχουμε, γιατί δεν είναι ε, πανεπιστημιακού, ακαδημαϊκού τύπου οι εκπαιδεύσεις αυτές. Εκπαιδεύσαμε πέρσι 29.000 αξιωματούχους και 90% από αυτούς δήλωσαν ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις ε, υπηρεσίες μας. Πάνω από 40% των δραστηριοτήτων μας αφοσιώνονται σε αυτήν την εκπαίδευση. Η κύρια έμφαση το 2018 ήταν για τη μετώπιση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος ε, αντιτρομοκρατία και αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευσης. Συχνά παρέχουμε την υπηρεσία αυτή της χώρες μέλη αλλά δεν ταιριάζει άμεσα με, τις, με τη ζήτηση. Εφόσον πρόκειται για συλλογή πληροφοριών, οι χώρες μέλη μας ζητούν και μέσω των υπηρεσιών τους συνεργασία. Οι δραστηριότητες που βλέπετε στην διαφάνεια ήταν επιτυχής και με πάρα πολύ στενή συνεργασία με Ευρωπόλ, Eurojust και Frontex για να περιλάβουμε και τη δική τους τεχνογνωσία στις ε, έρευνές μας. Ευχαρίστω σας παρουσιάζω τα πρώτα πορίσματα της αξιολόγησης που κάνουμε για τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την τροποποίηση της εντολής μας του 2016 μας επιτρέψατε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ανάγκες. έχουμε την ε, βάση σε επιστημονικά δεδομένα για τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες. Έως τώρα σε ορισμένους τομείς διαθέταμε κάποιες προφορίες, δεν είχαμε όμως ποτέ συνολική επισκόπηση, δηλαδή που θα πρέπει να διαθέσει τους πόρους για την εκπαίδευση των δυνάμεων επιβολής του νόμου η Ευρώπη στο μέλλον. Αυτό τώρα βάσει τη νέα μα συντολή μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Αυτό που κάναμε πρώτα ήταν να δούμε ποιε είναι οι βασικέ στρατηγικέ απειλέ για την Ευρώπη και μετά να εξετάσουμε πώ η κοινότητα των αρχών επιβολή του νόμου μπορεί να αντιμετωπίσει τι ε, απειλέ αυτέ. Ποιο είναι ο συγκεκριμένο ρόλο των ε, εταίρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθούν τα κενά που ενδεχομένω υπάρχουν. Βλέπετε για, σε ό,τι αφορά τον φόρτο εργασία, ποιε είναι οι δραστηριότητε και οι τομεί που έχουμε εντοπίσει. Στην άσκηση αυτή ρωτήσαμε 500 ειδικού από τις διάφορες υπηρεσίες χωρών μελών και διάφορους οργανισμούς για να διδαχθούμε από αυτούς για τα, ποια, θα, θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. Στην διαφάνεια αυτή μπορείτε να δείτε μια σύντομη επισκόπηση των βασικών δεδομένων που έχουμε ε, δει, ποιε είναι δηλαδή οι τα βασικά κενά των ικανοτήτων για να περιληφθούν στη μελλοντική δόμησή μας. Βλέπετε συλλογή προφοριών από ανοιχτέ πηγές, ε, χρηματοπιστωτικές έρευνες, άλλα στοιχεία, ε, παραχάραξη εγγράφων κλπ. Τα βλέπετε στη διαφάνεια. Οτιδήποτε έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια και τη σχετική τεχνολογία, ψηφιακές ε, προκλήσεις δηλαδή, αυτά βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Και αυτά θα αποτελέσουν και τη μελλοντική αλλαγή υποδείγματος. Πρέπει δηλαδή να ρίξουμε όλο το βάρος στην διαβίου κατάρτιση, των ε, προσώπων που ε, ε, συναποτελούν τις κοινότητες επιβολής του νόμου. Δεν μπαίνουμε υπερβολικά σε λεπτομέρειες, σας δείχνουμε όμως μια επισκόπηση των προτεραιοτήτων που έχουν σημειώσει για μας οι χώρες μέλη σε σειρά προτεραιότητας. Πρώτα για, τη, για θέματα διευκόλυνσης παράνομης μετανάστευσης, αντιτρομοκρατία, ε, σωματεμπορία, κυβερνοέγκλημα και ούτε καταξής. Δεν θα σας τα πω όλα, αλλά τα δεδομένα μας δείχνουν πλέον τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον για να υποστηρίξουμε αυτές τις κοινότητες επιβολής του νόμου στο μέλλον στην Ευρώπη σε μια στέρεα βάση για το σχεδιασμό των, επόμενων, των δραστηριοτήτων μάλλον των επόμενων ετών. Η επόμενη διαφάνεια τώρα ευχαρίστω να σας εξηγήσω ότι το 2018 όπως και τα προηγούμενα χρόνια ο οργανισμός σύμφωνα και με την εντολή του έχει αναλάβει και δραστηριότητε δημιουργία δεξιοτήτων και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα project για αντιτρομοκρατία με χώρε τη Εγγύης Ανατολή, ένα πακέτο για τη δυνατότητα χρηματοπιστωτικών ερευνών στην περιοχή των Βαλκανίων. Είναι πολύ σημαντικός ο σύνδεσμος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Και αυτό είναι προφανές, τουλάχιστον έγινε προφανές τα τελευταία χρόνια. Αυτό που κάναμε έως τώρα και είναι ένα ε, καλό εργαλείο για την συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Επιζητούμε διαρκή συνεργασία με τους ε, εταίρους μας στις δικαιούχους χώρες και αναζητούμε τη συνέργεια με όλους τους εταίρους εδώ και εκτός Ένωσης. Τονίζουμε πάντως όταν πηγαίνουμε στις χώρες αυτές εκτός Ένωσης και αυτό βεβαίως είναι αδιαμφισβήτητο και διαπρομάτευτο η τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αυτά είναι τα δύο αδιαπραγμάτευτα στοιχεία. Για αυτές τις ε, δραστηριότητες capacity building έχουμε συνεργασία και με άλλους εταίρους, βλέπετε ορισμένους όπως Ευρωπόλ, Frontex, EU, LISA και Eurojust, οι οποίοι όλοι αυτοί οι οργανισμοί συμμετέχουν πάρα πολύ στενά. Συνεργαζόμαστε επίσης και με Ευρωπόλ και η UNODC. Άλλα σημαντικά πορίσματα από το 2018 που είναι πολύ σημαντικά και για σας νομίζω. Το διαχειριστικό μας μοντέλο έχει περάσει και έχει πιστοποιηθεί ε, με ISO 9001 για το πώς δηλαδή ε, λειτουργούμε ε, και υπακούμε στα ε, βιομηχανικά πρότυπα, πρότυπα. Θέλουμε να προχωρήσουμε και σε επιστοποίηση ISO και για τις ε, εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Για το 2018 έχουμε εκτελέσει το 98% του προϋπολογισμού μας στο επίπεδο των υποχρώσεων και με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω ότι το ισχυρό σημείο του οργανισμού μας είναι μια απόλυτα στρατευμένη ομάδα με η οποία μας έπρεπε να επιτύχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τονίζω επίσης ότι δυστυχώς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις περικοπές μισθών και μισθολογίου στην Ουγγαρία. Αποτελεί πρόκληση αυτό για μας και ελπίζω ότι θα μπορέσει να διορθωθεί στο μέλλον. Η επόμενη διαφάνεια. Έρχομαι τώρα στο πρόγραμμα εργασιών του 2019. Θα ήθελα να το βάσω τώρα στο πλαίσιο και των διατηθειμένων κονδυλίων που θα το βρείτε στη δεξιά στήλη του ε, γραφήματος μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια έως 9,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τώρα και πρόσθετα κονδύλια τα οποία προέρχονται από τα project τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτό που θέλουμε τώρα να επιτύχουμε για το 2019 είναι να συνεχίσουμε πρώτα την αξιολόγηση των αναγκών στρατηγικής εκπαίδευσης αφενός μέσα σε μια πολυετή προοπτική η οποία θα πρέπει μετά να μετερμηνευτεί στην ε, κατέτος αξιολόγηση. Θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με τους εταίρους οργανισμούς στον τομέα αυτό και όπως είπα πριν θα συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους δικαιούχους αυτό είναι το core business, ο βασικός, η βασική μας δραστηριότητα. Το χαρτοφυλάκιο εκπαιδεύσεων προσφέρεται στις χώρες μέλη, όπου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς πολιτικές που είναι το κυβερνοέγκλημα, το έγκλημα το οποίο διευκολύνεται από μέσα στον κυβερνοχώρο και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία εκεί, σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας. Πέρσι θα φτιάξαμε και το κέντρο γνώσης σε πόλ αντιτρομοκρατίας με τους Ολλανδούς εταίρους μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία πάντα μέσα στα πλαίσια της στήριξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και προετοιμαζόμαστε και για τις αναφιόμενες ανάγκες Εκπαίδευση διότι πολλά πράγματα αναμένουμε να μας απασχολήσουν τα αμέσω επόμενα έτη. Προετοιμαζόμαστε και για τον νέο μας ρόλο όταν θα λειτουργήσει το νέο σύστημα ηλεκτρονικής τεχνολογίας, πληροφορικής, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και τις δραστηριότητες των χωρών μελών. Επόμενη διαφάνεια. Μίλησα πριν για την εξωτερική διάσταση της ε, ευρωπαϊκής ασφάλειας και αυτό που θα κάνουμε στο μέλλον είναι αφενός θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες και αποστολές ΚΕΠΑ, σε τρίτες χώρες δηλαδή, προετοιμασία των αποστολών αλλά και με άλλες δραστηριότητες και το κέντρο γνώσης πόλ όπου εκεί ηγούνται οι Πορτογάλοι εταίροι μας και επίσης για την συνεργασία με τρίτες χώρες όπως της Εγγύης Ανατολή και τη Βόρεια Αφρικής καθώς και των Δυτικών Βαλκανίων. Επιπροσθέτως θα εγκύπτουμε και σε θέματα ηγεσία και δεξιοτήτων γλωσσών, γλωσσικών δεξιοτήτων δηλαδή που είναι αναγκαία για την επιτυχή συνεργασία και είμαστε πεπισμένοι επίσης ότι για τη διεθνή συνεργασία και μέσα στην Ευρώπη χρειάζονται και στοιχεία στην εκπαίδευση δηλαδή, ηγετικών ικανοτήτων, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τι σημαίνει η βελτίωση της συνεργασίας μέσα στην Ευρώπη με τα υφιστάμενα εργαλεία. Θα θέλαμε επίσης να προωθήσουμε να, να, χρησιμοποιήσουμε μάλλον προωθημένες μεθοδολογίες εκπαιδεύσεως και να συμμετάσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην έρευνα διότι είμαστε πεπισμένοι ότι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες δυνατές γνώσεις που μπορεί να προσφέρει ο πανεπιστημιακός τομέας. Εδώ έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων που θα προσφέρουμε στις χώρες μέλη. Θα έχουμε συμμετοχή περίπου 30.000 συμμετεχόντων έχουμε 79 σεμινάρια μέσω του διαδικτύου, το λεγόμενο webinar, 100 residential activities, έχουμε 12 επιγραμμικές σειρές μαθημάτων και 6 ε, ενότητες, επιγραμμικές ενότητες και 330 προγράμματα ανταλλαγής όπως ε, με τον έρασμο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες να εργαστούν επί τόπου, hands-on, να συμμετάσχουν δηλαδή στις δραστηριότητες των εταίρων μας σημαντικό για τη μελλοντική συνεργασία. Πάλι για το 2019 θα έχουμε τη δεύτερη ομάδα σπουδαστών από το πρόγραμμα Master, JMP για πρόσωπα τα οποία θα καταλάβουν ηγετικές θέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις των χωρών μελών. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα με το οποίο, στο οποίο προβλέπεται συνεργασία με χώρες της Ανατολής και των Δυτικών Βαλκανίων, Βαλκανίων. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τις πιστοποίησεις 9001 και 29993 και κάτι νέο για φέτος. Έχουμε την πρόθεση να ανοίξουμε εκπαιδευτική ακαδημία στη Βουδαπέστη, σε European Cybercrime Training Academy, διότι θεωρούμε ότι οι προκλήσεις αυτές χρειάζονται κινητοποίηση όλων των δυνατοτήτων και πόρων των χωρών μελών, διότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Μιλώ για την κυβερνοασφάλεια. Ελπίζω ότι η Ακαδημία που σας ανέφερα θα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο. Ελπίζω να μην σας έφαγα πολύ χρόνο και είμαι στη διάθεσή σα αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανεί που θα ήθελε να θέσει ερωτήσει στον κύριο Σρόιντερ. Σας ευχαριστώ. Ορίστε, πρώτα όμως η Μπίργκιτ. Ευχαριστώ πολύ. Α, okay. <laughs> Είμαι βεβαίο ότι όλοι σας παρακολούθησαν προσεκτικά και γι' αυτό σήκωσαν το δάχτυλο για να κάνουν ερωτήσεις. Μία ερώτηση τυπικού χαρακτήρα. Είπατε ότι μέχρι τώρα 29.000 αξιωματούχοι πέρασαν από τις εκπαιδεύσεις σας. Αυτό ηχεί ως πολύ μεγάλος αριθμός. Από την άλλη μεριά, εάν κοιτάξω, οι αστυνομικοί στη Γερμανία είναι σε τριψήφιους αριθμούς και μόνο ένα συνδικάτο στην Γερμανία εκπροσωπεί 15.000 ε, ε, αστυνομικούς. Άρα τελικώς αυτοί 29.000 δεν μου φαίνονται τόσο πολύ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, έχετε κάποια επιρροή σχετικά με το ποιος προσέρχεται τις εκπαιδεύσεις αυτές και εκ του αντιστρόφου θα προσπαθήσετε να φτάσετε να μπορέσετε δηλαδή να εκπαιδεύσετε ε, αξιωματούχους της αστυνομία και των άλλων αρχών επιβολής του νόμου που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα τα οποία πρέπει να εκπληρώσετε και τα οποία θα έχετε και στο μέλλον, το ερώτημα που τίθεται επιπροσθέτως είναι με όλη αυτή την δέσμευση αλλά και με τα χρήματα που δαπανώνται και θα δαπανηθούν και στο μέλλον. Ποια η υποστήριξη δίνεται στις ίδιες τις χώρες μέλη ώστε να συνεχίσουν τις εκπαιδεύσεις αυτές, να τις εμβαθύνουν, να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν και άλλους αστυνομικούς, γιατί βεβαίως τα όσα κάνει ο οργανισμός σας σε πολ δεν, αρκεί, δεν αρκούν. Και βλέποντας τώρα και τις σειρέ προτεραιοτήτων με τις οποίες, ε, με τις οποίες ασχολείστε Βλέπω ότι ο κατάλογος αυτός θα υπάρχει τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία ως έχει. Ή θεωρείτε ότι μπορούν οι προτεραιότητες αυτές και να ανατραπούν ε, αναλόγως των εξελίξεων. Πώς το βλέπετε. Ο κύριος Ντεπρέ ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σχόλιο όσον αφορά την παρουσίαση. Την εξετίμησα πολύ. Υπήρξε σαφέστατη. Και είπα στον εαυτό μου βλέποντας την παρουσίαση ότι σύντομα θα φτάσουμε σε κινούμενα σχέδια. Τόσο πιο σαφής ε, γίνεται η απεικόνηση. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως της παρέμβασης. Όπως είπε η κυρία Σίπελ, 29.000 ε, αξιωματικοί αστυνομία εκπαιδεύονται. Από πού προέρχονται, από τα κράτη-μέλη κανονικά. Κάποια κράτη-μέλη ε, απευθύνονται περισσότερο σε εσά και κάποια κράτη-μέλη καθόλου. Ίσως κάποιοι χρειάζονται ή αξίζουν να εκπαιδευτούν περισσότερο και δεν είναι εκεί. Έχετε κάποια ιδέα, κάποια εικόνα. Καταρτίζεται αυτός που είναι ήδη καταρτισμένοι ή αστυνομικού που πραγματικά χρειάζονται βελτίωση όσον αφορά την κατάρτισή του. Μετά, αυτή την εβδομάδα συνάντησα τη νέα διευθύντρια της Europol και μου είπε ότι θα πάει στα διάφορα κράτη-μέλη. Και έκανε, πήγε στα διάφορα κράτη-μέλη μάλλον και κατέληξε ο συμπέρασμα μετά την επίσκεψή της ότι σε δύο τομείς η Europol πρέπει να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό της και το έργο της. Το αναφέρατε πρώτα απ' όλα στην οικονομική, στο οικονομικό έγκλημα, στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος. Και μετά στα ναρκωτικά. Για την ώρα τα ναρκωτικά πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αυξάνεται καθημερινά. Όλο και περισσότερο βλέπουμε σκληρά ναρκωτικά. Δεν μιλάμε για την κάναβη. Σκληρά ναρκωτικά που μπαίνουν στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Έχει συγκεκριμένε πληροφορίε. Όσον αφορά τον εντοπισμό των ναρκωτικών, τι βέλτιστε πρακτικέ, συντονίζεστε με τη Europol. Όσον αφορά τι προτεραιότητε, διότι μου είπε ότι είναι δύο από τι προτεραιότητε ε, στις οποίες θα επενδύσει πολύ τα επόμενα χρόνια. Η Σοφίντφελτ, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σρέντερ για την ε, παρουσίασή σας. Ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνατε. Εξεπλάγιν πρέπει να πω καταρχάς και ανησύχησα τον άκουσα αυτό που είπατε προς το τέλος. Ότι έχετε πρόβλημα να προσελκύσετε προσωπικό ε, στη Βουδαπέστη. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται διευκρίνηση. Μάλιστα διότι ήταν επίμαχο ζήτημα η επίλεξη της έδρας την εποχή εκείνη. Πέρα από τα σημαντικότατα θέματα που ήδη αναφέρθηκαν και τις ερωτήσεις που απευθύνθησαν, αν δούμε τα εγκλήματα τα οποία εξηχνιάζεται και εξετάζεται είναι, σε, είναι το κυβέρνο έγκλημα, η τρομοκρατία, απόμακρα από τον απλό άνθρωπο. Είχαμε επαφή διαλληλογραφίας επί σειρά ετών για διάφορα θέματα και για προβλήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων όπως η οικιακή βία 2.500 νεκρούς ε, κάθε χρόνο έχουμε στην Ευρώπη. 2.500. Αν το συγκρίνεται αυτό με, τα, με τους νεκρούς που είναι θύματα τρομοκρατίας, θα έλεγα ότι υπάρχει κάθε λόγος να αναβαθμίσουμε την οικιακή βία σαν προτεραιότητα στο έργο σας. Θα πείτε ίσως ότι αυτό είναι πολύ τοπικό πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είναι γενικό πρόβλημα και είναι κάτι που καλύπτεται την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν δείτε την οδηγία για τα θύματα, έχουμε προγράμματα κατά της έμφυλης βίας κλπ. Έχετε κάθε λόγο λοιπόν να παράσχετε κάποια κατάρτιση σε αυτό το τομέα. Συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κ. Δεπρέ. Πιθανότατα ίσως να καταρτίζετε κάποιους αστυνομικούς από χώρε όπου ήδη έχουν πολλή κατάρτιση αλλά και για συγκεκριμένους τομείς αστυνόμευσης. Κάποιους τομείς ε, στους οποίους, ε, για τους οποίους οι αστυνομικοί λένε αυτό είναι θέμα ιδιωτικό. Μιλάμε για ενδυμική βία που στρέφεται κυρίως κατά των γυναικών. γυναικών συγγνώμη. Το ίδιο για τους ΛΟΑΔ και τα διεμφυλικά άτομα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο διάκριση αλλά και βία. Και βία και από τους αστυνομικούς. Το ίδιο για τους ε, εργαζόμενους στον τομέα των σεξουαλικών υπηρεσιών. Είπατε καθήκον της ΕΠΟΛ είναι να καταρτήσει, να θεσπίσει κάποιους διοντολογικούς κανόνες. Και αυτά που ανέφερα είναι σημαντικά να ληφθούν υπόψη. Αναφερθήκατε και στην κακομεταχείριση των παιδιών αλλά κυρίως στο ίντερνετ. Αλλά υπάρχει μεγάλη κακομεταχείριση, μεγάλο ποσοστό κακομεταχείριση στον πραγματικό κόσμο. Αλλά είναι πιο δύσκολο αυτό. Πολύ πιο εύκολο να κάθεται κανείς, εύκολο τέλο πάντων, τρόπος του λέγει. Δεν θέλω να το πω έτσι. Ε, αλλά θα πρέπει να εστιαστούμε επί τη κακομεταχείρισης των παιδιών στον πραγματικό κόσμο, όχι μόνο στο διαδίκτυο. Συνεργαστήκατε με διάφορου φορεί, αλλά λείπουν δύο. ΦΡΑΜ και το EIGE που είναι η υπηρεσία για την ισότητα των φύλων. Δεν αναφέρατε αυτούς τους φορείς. Ευχαριστώ, Σοφή. Ο λόγος και πάλι στον κύριο Σρέντερ. Thank you very much and thank you really. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και ποιοι συμμετέχουν και αν όντως καταρτίζουμε τους κατάλληλους. Όπως σας προσπάθησα να σας εξηγήσω, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το επιχειρησιακό μας μοντέλο και να δούμε ακριβώς ε, για ποια θέματα χρειάζεται κατάρτιση και εκπαίδευση και να δούμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να έχουμε σωστές ομάδες στόχους. Αυτό επιχειρήσαμε εμείς στη ΣΕΠΟΛ, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία και με τους εταίρους μας σε εθνικό επίπεδο. Ε, αυτοί έχουν δική τους εντολή και εντοπίζουν σε εθνικό επίπεδο ποιοι είναι οι κατάλληλοι και χρήζουν κατάρτιση και εκπαίδευση για να του στείλουν στι δικέ μα δραστηριότητε, ώστε οι εθνικέ αρχέ συναρμόδιε να στέλνουν του κατάλληλου. Επίση, έχουμε βελτιώσει το σύστημα τα τελευταία χρόνια, ώστε όντω ε, να συμμετέχουν οι κατάλληλοι στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μερικέ φορέ, μάλιστα, έχουμε πολύ περισσότερου ε, εθελοντέ από ότι θέσει στι ε, εκπαιδεύσει και τι καταρτήσει μα. Ακόμη και μεγάλους εταίρους δίνουμε συνήθως ε, μια θέση ανά χώρα μέλος, γιατί δεν έχουμε και πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, οπότε πρέπει να περιορίσουμε τη θέση. Και ο ένας ε, υποψήφιος ανά μέλος μπορεί να ικανοποιεί τις μικρές χώρες, αλλά για μεγάλες χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Και ε, δεν αρκούν τα σεμινάρια που κάνουμε στην έδρα μας. Γι' αυτό και προσπαθούμε να επεκτείνουμε την κατάρτιση σε online μαθήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχει περιορισμό θέσεων. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα και γλωσσικό. Μερικοί δεν συμμετέχουν στι δραστηριότητέ μα, γιατί κυρίω γίνονται στα αγγλικά τα σεμινάρια. Θα πρέπει ίσω κάτι να γίνει εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο αντικτύπο. Αλλά αυτό θα πρέπει να το ε, εξετάσουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει επίση μια πρόοδος ε, καθορίζουμε τις δραστηριότητες και τις ομάδες στόχους. Ποιος είναι ο κατάλληλος για κάθε δραστηριότητα, είτε σε αίθουσα είτε στα μαθήματα γενικώ. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση έχει βελτιωθεί για να πιάνουν το στόπο τα μαθήματα που δίνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, ε, για να κρατήσουμε ένα συνεχή αντίκτυπο και επιπτώσει στα κράτη-μέλη. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε και τους εκπαιδευτές ε, ώστε να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και ωφέλεια των σεμιναρίων. Επίσης έχουμε και πρόγραμμα ανταλλαγής της ΣΕΠΟΛ. Ένα τμήμα του προγράμματος ε, ε, δεν επιτρέπει μόνο την μετακίνηση από το α στο β σημείο. Όλοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια για το τι θα κάνουμε την επιστροφή, μετά την επιστροφή τους, μετά την επίσκεψή τους δηλαδή, τι συνέχεια θα δώσουν δεν είμαι αφελής, δεν γίνονται όλα τέλεια, αλλά είχαμε πολλά καλά παραδείγματα, ώστε πραγματικά ε, όσοι υποφελήθηκαν από τα προγράμματα ανταλλαγής, στη συνέχεια μετέδωσαν αυτές τις γνώσεις ε, και στους συναδέλφους τους ε, στη χώρα τους. Επίσης, θα πρέπει και τα κρατημέλη να συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες μετάδοσης των γνώσεων των σεμιναρίων. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, ε, με βάση τις συνεντεύξεις που είχαμε τελευταία διετία σας δώσαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σίγουρα οι απειλές ε, και ε, οι προκλήσεις εξελίσσονται και θα πρέπει να τις παρακολουθούμε. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δώσαμε, διαπιστώσαμε ότι η μετανάστευση είναι από, από τα σημαντικότερα ζητήματα. Για κάποιε χώρε η μεταναστευτική πίεση δεν είναι τόσο υψηλή όσο στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα. Απλώ αλλάζει η σειρά των προτεραιοτήτων. Επίση, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο κατάλληλο μηχανισμό εδώ. Πάντω, χαίρομαι που για πρώτη φορά σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλε τι υπηρεσίε είχαμε μια πολύ καλή επισκόπηση. Βέβαια, γνωρίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί επιφυλακτικοί, γιατί δεν ξέρουμε τι πρόκληση θα ανακύψει του χρόνου, τι καινούργια απειλή. Ελπίζω η τρομοκρατία να μην είναι τόσο σημαντική απειλή όπως στο παρελθόν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου, του, του παραχρόνου. Ο κύριος Ντεπρέ μίλησε για τον υψηλό αριθμό και πώς γίνεται η διαφοροποίηση εντός των ομάδων στόχου. 29.000 ε, ήταν όσοι υποφελήθηκαν. Από μόνος του αριθμός είναι σημαντικός, αλλά είναι 1,1 ουσιαστικά των αρχών ε, των συμμετεχόντων στις αρχές επιβολής του νόμου. Εμείς βλέπουμε πού θα πρέπει να στηρίξουν τα κοινοτικά κονδύλια της ομάδες της αρχές επιβολής του νόμου. Επίσης, έχουμε και το θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Προσπαθούμε έτσι να συνδυάσουμε τις διάφορες, τα διάφορα επίπεδα και να είμαστε πιο επιτυχημένοι στο μέλλον. Επίσης, προσπαθήσαμε να καθορίσουμε ε, καλύτερα τις ομάδες στόχους για να δούμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι που θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεδομένης η διαφορά στις δομές των κρατών μελών είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Πάντως ευτυχώ μέχρι ε, το 2016 είχαμε μια διευρυμένη εντολή Πάντως, ό,τι αφορά τι στάσει τι πληθυσμιακέ, θα ήθελα περισσότερη ανάμειξη και των τελωνιακών υπαλλήλων. Ε, συνήθως έχουμε αστυνομικού που συμμετέχουν, αλλά από άλλα επαγγέλματα έχουμε κάποιου δικαστέ λίγου αγγελείς, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να επεκτείνουμε τα σεμινάρια και την εκπαίδευση και σε άλλου υπαλλήλου. Επίση, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε ε, παντού ή σε όλους όπως θα θέλαμε. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το έπακρο τα ηλεκτρονικά εργαλεία, γιατί ε, είναι πολύ πιο μεγάλες οι δυνατότητες από ότι το μάθημα στην αίθουσα. Και επειδή με τους πόρους τους λίγους που έχουμε δεν μπορούμε να φτάσουμε σε όλους. Τώρα, αν εκπαιδεύουμε τους κατάλληλους ε, ανθρώπους. Όπως σας είπα γενικώ θεωρούμε ότι έχουμε ένα σωστό και κατάλληλο δείγμα. Όχι αρκετούς βέβαια όπως σας είπα, έχουμε τριπλάσιους αριθμών υποψηφίων από τις θέσεις πολλές φορές σε κάποια σεμινάρια. Φυσικά θα θέλαμε να εκπαιδεύσουμε πολύ, πολύ περισσότερους, αλλά δεν έχουμε αρκετούς πόρους αυτή τη στιγμή. Επίσης, ρωτήσατε αν λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες της Europol. Ναι, έχουμε θαυμάσια σχέση με την Europol και με τον εκτελεστικό διευθυντή. Οικονομικό έγκλημα. Γνωρίζω ότι το διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα είναι σημαντικό φαινόμενο και επίσης θα πρέπει να ανακτήσουμε τα κονδύλια, ε, να, κάνουμε, να βελτιώσουμε τις έρευνες και να δούμε πού έχουν εκτραπεί αυτά τα κονδύλια. Επίσης, όπως σας είπα στο σχέδιο με τα Δυτικά Βαλκάνια, επικεντρωθήκαμε κυρίως σε οικονομικές ε, ερευνήσεις απατών. Και για τα ναρκωτικά επίσης χρήζει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να βρούμε, να εντοπίσουμε τα παράνομα εργαστήρια, να τα διαλύσουμε γίνεται, να εξαρθρώσουμε τέτοια κυκλώματα. Άλλωστε το, τα ναρκωτικά είναι παγκόσμια πρόκληση και στο μέλλον θα γίνει σωστό πιο οξύ πρόβλημα και στην Ευρώπη. Ε, βλέπουμε τα στοιχεία από άλλες περιοχές του κόσμου και αν τα προβλήματα αυτά μετακινηθούν και προς την Ευρώπη θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα γιατί σε κάποια θέματα της αγοράς ε, των ναρκωτικών. Μερικές φορές δεν εισάγουμε μόνο ναρκωτικά, αλλά και εξάγουμε. Το σύστημα είναι διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν. Ε, συντονισμός με τη Europol. Όπως σας είπα, είναι εξαιρετική η συνεργασία με τη Europol και στο σχέδιο δράσης μας βλέπουμε σε ποιες δραστηριότητες η Europol έχει καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη και όπου μπορούμε στηρίζουμε την Europol με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων για τον κύκλο πολιτική, για παράδειγμα. Επίση, έχουμε σε όλε τι ομάδε και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα κατάρτιση για, να, για τα θέματα πολιτικής, ώστε αυτές οι ομάδες να είναι πιο αποτελεσματικές χάρη σε αυτή την εκπαίδευση που προσφέρουμε. Επίσης, από αναλυτικές μελέτες ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, είναι θετικές οι μελέτες και δείχνουν ότι οι υπηρεσίες ε, που δίνει σε πόλ για τις δραστηριότητες αντικτύπου είναι πολύ θετικές και έχουν πολύ καλό αντικτύπο. Τώρα για το ποιους προσελκύουμε. Μέχρι στιγμής η πρόκληση, κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι η έδρα στη Βουδαπέστη, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ε, η Βουδαπέστη είναι μια χαρά πόλη και το λέω από προσωπική εμπειρία γιατί εκεί ζω. Βέβαια, ο, ο, ο διορθωτικός συντελεστής είναι πρόβλημα γιατί είναι δύσκολο να βρούμε εξειδικευμένο προσωπικό στη συγκεκριμένη αγορά και έχουμε και άλλες ε, ε υπηρεσίες ε, και οργανισμούς που βρίσκονται στις κάτω χώρες ή αλλού. Εκεί ο συντελεστής δεν είναι και πολύ ελκυστικός ο διορθωτικός. Πάντως έχουμε εξαιρετικό προσωπικό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ε, ο αριθμός ε, αιτήσεων για εργασία στη ΕΠΟΛ. Γιατί σίγουρα ε, το μισθολογικό επίπεδο περι, περιμένουν οι υποψήφοι από τις δυτικές χώρες, κυρίως της Ευρώπης, είναι υψηλότερο από αυτό που προσφέρουμε στη ΣΕΠΟΛ. Σε ό,τι αφορά την ενδογενειακή βία, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα εδώ και πολλά χρόνια και σίγουρα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη μας λένε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικότερες προτεραιότητες τα οποία ζητούν τη συνεργασία μας. Και εκεί γίνεται διάκριση των διαφόρων ε, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς σε ενωσιακό επίπεδο, σε κοινωτικό επίπεδο και τι θα πρέπει να καλυφθεί σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αρκούν οι δικές του δραστηριότητε για την ενδοοικογενειακή βία και εμεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλα θέματα. Δεν θέλω να κρίνω αν αυτό ισχύει ή όχι αλλά σεβόμαστε την ε, γνώμη των κρατών μελών που λένε ότι αρκεί η δική τους δράση για την ενδοοικογενειακή βία. Επίσης ε, και για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ μας, μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματά τους. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τα εγκλήματα εις βάρος τους, τα εγκλήματα μίσους γενικώ και μεσαλλοδοξίας. Αλλά έχουμε πολλές δραστηριότητες. Δεν έχουμε ειδική δραστηριότητα για το θέμα αυτό. Προσπαθούμε να εντάξουμε αυτή τη διάσταση προστασία των ΛΟΑΔ σε άλλες δραστηριότητες. Επίσης έχουμε και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, άλλες, ε, και άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες με τις οποίες έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία. Επίσης, ε, στις τρίτες χώρες ε, προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τη δική μας αντίληψη, την ευρωπαϊκή αντίληψη για τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το δούμε μονομένα, αλλά στα, ζητήματα, στα γενικά ζητήματα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην καταπολέμηση των δεκτύων των ε, εγκλημάτων μίσους. Επίσης, για τις ιερόδουλες, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και προσπάθησα να το εξηγήσω και προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με εσάς και με άλλους εταίρους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, πώς να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας, αλλά είναι και θέμα εθνικό εδώ και θα πρέπει και τα κρατη να συνεργαστούν και να μας στηρίξουν. Ευχαριστώ κύριε Σρέντερ. Um, Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Καλή επιστροφή στη υπέροχη Βουδαπέστη. Συμφωνώ. Υπέροχη, πολύ ωραία πόλη. Πάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, όπου θα προεδρεύσω του εαυτού μου. Οπότε κάποιος θα στιμάσει το χρονόμετρο, διότι νομίζω ότι αυτό θα ήταν δίκιο. Διότι πάμε τώρα στην εξέταση τροπολογιών που έχουν υποβληθεί όσον αφορά την πρόταση για αναδιατύπωση της οδηγίας περιπιστροφών του 2010. Ε, εγώ 120 τροπολογίες υπέβαλα σαν συνεισηγήτρια και οι άλλοι σκιώδεις άλλε 534 τροπολογίες, σύνολο 654 τροπολογίες. Να σας πω ποια είναι η κατάσταση. Γι' αυτό ήθελα να αρχίσετε το χρονόμετρο. Και μετά, αφού σας περιγράψω την όλη κατάσταση, θα στραφώ προς τους ε, σκιώδεις. Εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένη με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν την είχαν εξετάσει διεξοδικά. Τη έλειπε η αξιολόγηση αντικτύπου και αποφασίσαμε γι' αυτό σαν Επιτροπή να κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση αντικτύπου που παρουσιάστηκε και εδώ στην Επιτροπή πρόσφατα. Πέρα από αυτό, δεν ξέρω, 7-8 συνεδριάσεις των σκιωδών διοργανώσαμε και εκεί καλέσαμε τις οργανώσεις του ΟΙΕ, της κοινωνίας των πολιτών, αξιωματούχους που εργάζονται στον τομέα των επιστροφών, νομικούς, καλέσαμε πολλούς ειδικού για να σχηματίσουμε εικόνα του θέματος. Εάν θέλουμε μια πραγματικά αποτελεσματική διαδικασία επιστροφών που συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βάσει αυτών ξεκινήσαμε τις εργασίες και οι προτάσεις που επεξεργάζομαι εστιάζονται επί των εθελοντικών επιστροφών. Η αξιολόγηση αντικτύπου δείχνει ότι αν θέλει κανείς να αυξήσει τον αριθμό ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν διότι δεν έχουν τα κατάλληλα έγγραφα να παραμείνουν, πρέπει να εστιαστούμε επί εθελοντικών επιστροφών. Ενώ η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιαζόταν πιο πολύ στο να ε, προσπαθήσει κανείς από τα κέντρα κράτησης να επιστρέψει τους ανθρώπους αυτούς στις χώρες τους. Αυτό πιστεύω ότι είναι αντιπαραγωγικό, όχι ότι η κράτηση δεν μπορεί να συμβεί, διότι πρέπει να λαμβάνει η χώρα αυτό σαν ε, το τελευταίο μέσο που θα χρησιμοποιήσει. Δεν θα πρέπει να είναι όμως αυτό που έχει προτεραιότητα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν διαφορετικές ιδέες, λίγο διαφορετικές αλλά παρόμοιες. Το άρθρο Έξι πρέπει να επεξεργαστούμε ε, που αναφέρεται στις ε, παγωγές όπου ε, εξαφανίζονται οι άνθρωποι που δεν έχουν κατάλληλα έγγραφα φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα, παράτυπα, δεν έχουν δελτία ταυτότητας, δεν μπορεί αυτός που έρχεται να πληρώσει για να ζήσει, δεν έχει διεύθυνση αυτός ο άνθρωπος όπου μπορεί να μείνει. Αυτά είναι τέσσερα από τα κριτήρια αυτής της παράνομης διαμονής και εκεί ε, δεν βοηθούν οι πολιτικές ομάδες ε, να μας πούνε ποιος είναι ο κίνδυνος αυτοί οι άνθρωποι να ξεφύγουν και να παραμένουν χωρίς να έχουν εντοπιστεί παράνομα. Λοιπόν, λοιπόν, το να φοβάται κανείς ότι ο άνθρωπος αυτός θα ξεφύγει οδηγεί στο να συλλαμβάνεται εύκολα και να κρατείται και να μην ε, μπορεί να φύγει εθελοντικά και αν είναι να απομακρυνθεί ε, τελικά χωρίς τη βούλησή του άνθρωπος απαγορεύεται η είσοδος του στο μέλλον και έτσι δεν μπορεί ε, να αποφασίσει ελεύθερα αυτός ο άνθρωπος διαμένει παράνομα εάν θέλει να επιστρέψει, να επιλέξει να επιστρέψει. Λοιπόν, θέλουμε να διευκρινίσουμε και τα δικαιώματα των μεταναστών που πρέπει να επιστραφούν και τις υποχρεώσεις που έχουν οι αρχές να δώσουν τις κατάλληλες σωστές πληροφορίες στον άνθρωπο αυτό, στο μετανάστη. Μετά χρονοδιαγράμματα για ε, αναφέρεται αυτό σε διάφορα άρθρα και επειδή υπάρχουν πολλές αναφορές είναι δύσκολο να βγάλει άκριο ο μετανάστης για να μπορεί να υποβάλει την έφεση και είναι πολύ δύσκολο και αρχές να εφαρμόσουν τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή εφέσεων και πολλοί συνάδελφοι έχουν υποβάλει τροπολογίες ούτω ώστε τελικά να είναι πιο εύλογο το χρονοδιάγραμμα που ε, προτείνεται. Υπάρχει διαδικασία μεθοριακή που προτείνεται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωπικά εγώ τα φέρα σε την τροπολογία μου και βλέπω διάφορους συναδέλφους από διάφορες ε, πολιτικές ομάδες να κάνουν το ίδιο, διότι δεν υπάρχει ακόμα σαφήνεια όσον αφορά τις μεθοριακές διαδικασίες κατά την άφηξη, άρα δεν μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα στην άφηξη στα πλαίσια της οδηγίας επιστροφών. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέλω να αντιμετωπίσω. Να μην αναμίξουμε την κράτηση προς επιστροφή με την κράτηση εκείνων που έχουν ποινικό παρελθόν. Έχουν ποινικό μητρό. Δεν πρέπει να συναθρίζουμε, να βάζουμε στο ίδιο κέντρο κράτηση... σε αυτές δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνται πραγματικοί εγκληματίες ή που ίσως είναι τρομοκράτες θα πρέπει να ενταχθούν σε ποινικέ διαδικασίες και να επιστραφούν από μια κανονική φυλακή. Αν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε και βρίσκουμε μια διέξοδο αυτούς να τους βάλουμε σε κέντρα κρατήσεως μεταναστών, τότε φέρνουμε ανθρώπους που είναι στην εθνική κατάσταση μετανάστες που δεν έχουν κάποιο ποινικό μητρό σε επαφή με εκείνους που πραγματικά να τους θέσουν σε κίνδυνο. Και διευκολύνουμε τις αρχές μας να μην εξηχνιάσουν ποινικέ υποθέσει και να βρίσκουν την πιο εύκολη διαδικασία επιστροφή ενό συγκεκριμένου μετανάστη από το κέντρο κράτη μεταναστών. Αυτό δεν είναι επικοδομητικό και αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα, ποινικά δικήματα και στην επικράτειά μα και αλλού θα πρέπει να δικαστούν στην Ευρώπη, αν πρέπει να δικαστούν να δικάζονται. Δεν πρέπει να τους διευκολύνουμε. Αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα πρέπει να δικαστούν και ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ποινή που αφορά φυλάκιση και όχι κράτηση του κέντρα κράτησης μεταναστών. Πού είμαι τώρα από πλευράς χρόνου, τι άλλο έχω να πω. Λοιπόν, έχουμε συνεδρίαση των σκιωδών. Έχει προγραμματιστεί για 7 Μαρτίου και πριν από αυτή της 7ης Μαρτίου τη συνεδρίαση θα σας δώσω συμβαστικές τροπολογίες για να κουβεντιάσουμε κυρίως όσον αφορά τον κίνδυνο διαφυγής αυτών των παρανόμων μεταναστών, απαγόρευση επανεισόδου τους, ε, πώς οι εθνικές αρχέ θα πρέπει να είναι πιο δέκτικες όσο το μήνυμά μας, δηλαδή ότι το μέλλον είναι οι, οι επιστροφές και να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα. Ήδη την περασμένη εβδομάδα είχαμε συναντήσει σκιωδών, παρόλο που δεν είχαμε έτοιμε όλε τι μεταφράσει, διότι κατανοώ ότι ο χρόνο μα πιέζει και θέλουμε ένα αποτέλεσμα τη ΛΥΜΠΕ και ψηφοφορία ενδεχομένω στην Ολομέλεια πριν πάμε στι εκλογέ, στην προεκλογική εκστρατεία και στη διακοπή για τι εκλογέ. Αυτά έχω να πω ω εισηγήτρια. Α κουβεντιάσουμε τώρα. Α ακούσουμε του σκιώδει ο κύριος Κοέλιο εκπροσωπεί την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Άννα Μαρία πράγματι δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματι της στο ΕΛΚ καλωσορίζει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρηση της ισχύουσης ε, οδηγίας περί επιστροφών. Θέλουμε οι επιστροφές να είναι αποτελεσματικότερες ενώ θα εγγυόμεθα το σεβασμό των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων στις τροπολογίες μας θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες με συμφωνίες επανεισδοχής για να διευκολύνουμε την εθελοντική επιστροφή. Ταυτόχρονα θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τα μέτρα αναγκαστικής επιστροφής όταν απαραίτητο. Έχουμε πέντε προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, ο κίνδυνος διαφυγής των μεταναστών θεωρεί το ΕΛΚΟ ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατάλογο κριτηρίων που δεν θα είναι εξαντλητικός κατάλογος, ούτως ώστε να προσανατολίζουμε τα κράτη-μέλη για αξιολόγηση που ε, καθορίζει τον κίνδυνο διαφυγής αυτών. Δεν υποστηρίζουμε τη διαγραφή όλου του άρθρου, όπως προτείνει η συγγήτρια. Εξαλείφουμε τα πρώτα τρία κριτήρια αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον κατάλογο. Θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση το κάθε θέμα για να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια εξετάζοντας τη συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά κάθε μετανάστη ξεχωριστά. Δεύτερο, υποχρέωση συνεργασίας. Το ΕΛΚ υποστηρίζει διασύνδεση μεταξύ συνεργασίας και διαδικασιών που εφαρμόζονται. Το καθήκον συνεργασίας είναι σημαντικό επίσης για την αποφυγή διαφυγής και δευτερογενών μετακινήσεων. Τι συνέπειε μη συμμόρφωση με την υποχρέωση συνεργασίας θα, θα πρέπει να δέχεται ποινέ που θα είναι αναλογικές και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται η τύχη των παιδιών. Μετά η απαγόρευση εισόδου. Το ΕΛΚ υποστηρίζει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να εκδώσουν απαγόρευση εισόδου όταν αυτό ενδείκνεται σε περίπτωση παιδιών και σε περιπτώσεις θελοντικών επιστροφών θα πρέπει να είναι περιορισμένο αυτό το μέτρο. Τέταρτον, οι συνοριακές διαδικασίε, Το ΕΛΚ υποστηρίζει τη συμπερίληψη συγκεκριμένη διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόσει τα σύνορα. Θα επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική επιστροφή των μεταναστών που προφανώς δεν χρειάζονται διεθνή προστασία και που ήδη έχουν περάσει στα σύνορα από τη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου εξαιρούνται ευάλωτα άτομα όπως είναι τα παιδιά. Πέμπτο και τελικό σημείο. Τα δικαιώματα των παιδιών. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες μαζί με την ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών για να αυξηθεί η προστασία των παιδιών καθ' όλη τη διαδικασία της επιστροφής. Καταρχάς, η εξάλληψη της κράτησης για τα συνόδευτα παιδιά για οικογένειε με, τα οικογένειες παιδιά θα πρέπει να μπουν σε εναλλακτικέ εγκαταστάσεις, όχι σε κέντρα κράτηση. Τα παιδιά θα πρέπει να τύχουν νομική αρρωγή και οι κυδεμόνε των παιδιών θα πρέπει να ενημερώνονται και θα πρέπει οι πληροφορίες που δίνονται στο παιδί να δίνονται με φιλικό τρόπο. Και η επιστροφή να αναβάλλεται μέχρι τελειώσει το παιδί το σχολικό έτος και η μη συνεργασία ή η διαφυγή, η η περί διαφυγής θα πρέπει να ξερεί τα παιδιά γιατί δεν είναι υπεύθυνα για αυτές τις πράξεις. Πριν απόφαση περί επιστροφής που αφορά ένα παιδί, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα καλύτερα συμφέροντα του παιδιού εξετάζοντας μακροπρόθεσμες λύσεις για το παιδί και όταν λαμβάνεται απόφαση για επιστροφή να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιστροφή στη χώρα ε, καταγωγής. Η Άννα Μαρία ευχαριστεί την εισηγήτρια, την κυρία Σαρτζεντίνη και για την καρποφόρα συνεργασία και προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά αυτό το χαρτοφυλάκι. Ευχαριστώ. Η Σιλβή με έχει το λόγο. Ευχαριστώ και συνεχίζω εκεί που σταμάτησε ή τελείωσε ο Κάρλος Κοέλιο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την προσωρινή πρόοδο την κυρία Σαρχεντίνη για την αγαστή συνεργασία που είχαμε, αλλά και τους υπόλοιπους και οδησηγητές. Με την ε, μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας ε, έχουμε πραγματικά μία οδηγία που έχει ιστορία και αν θέλουμε να προσεγγίσουμε νυφάλια το κείμενο θα πρέπει να κρίνουμε ότι αν οι επιστροφές ε, καταστούν δυνατές θα πρέπει να είναι απόλυτα ισορροπημένες ό,τι αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. η ομάδα μου έχει ε, υποβάλλει καμιά εκατοσταριά τροπολογίες ε, για διάφορους τομείς. Θα τους αναφέρω εν συντομία με τυχαία σειρά. Η βασική μας προτεραιότητα είναι τα 11 μέσα, τα, το δικαίωμα προσφυγής. Προτείνουμε τουλάχιστον 15 μέρες για την κατάθεση ε, έφεσης απέναντι, απέναντι μιας απόφασης επιστροφής, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ημέρη προθεσμία και θέλουμε επίση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Δεύτερο, για την κράτηση. Προτείναμε μείωση τη κράτησης, της περίοδου κράτηση, που ήταν 18, δηλαδή 6 δύο φορέ ανανεώσιμη. Εμεί προτείναμε δύο μήνε προθεσμία και να επιτρέπεται ανανέωση μόνο δύο φορέ για τη διάρκεια της κράτησης. Επίσης, τα κείμενα είναι σαφέστατα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση ε, της ε, διάρκειας αυτής για άτομα που δημιουργούν κίνδυνο στη δημόσια ασφάλεια, εννοείται. Για το άρθρο 20, κράτηση ανηλίκων. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που ε, έχουμε ανηλικούς θα πρέπει να απογορευτεί η κράτηση των ανηλίκων, η κράτηση ε, οικογενειών. Τέταρτος θέμα, ο κίνδυνος διαφυγής απόδραση ή Το άρθρο 6 που προσδιορίζει αυτό τον κίνδυνο της διαφυγής ε, περιλαμβάνει ένα μη εξαντλητικό κατάλογο, έναν ενδεικτικό κατάλογο με πολύ ε, ευρεία κριτήρια. Εσείς αποφασίσατε να καταργήσετε αυτό τον κατάλογο και να κρατήσετε το κείμενο της προηγούμενης οδηγίας. Άρα τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν ή να διατηρήσουν τα δικά τους κριτήρια. Επίσης, προτείνεται να έχουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο, αν είναι να κρατήσουμε κατάλογο, με σαφή κριτήρια, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ερμηνείας ή να περιορίσουμε το, το περιθώριο ερμηνείας. Να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε ώστε να αποφύγουμε να υπάρχουν ακατάλληλα κριτήρια από κάποια κράτη-μέλη όπως ε, την έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων που χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο από κάποια κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά επίσης την διαχείριση αυτών των επιστροφών, μια προτεραιότητα μας είναι να καταργηθεί παράγραφος, το δάφιο της παραγράφου 14 που ζητούσε την δημιουργία νέας βάσης δεδομένων σε σχέση με τον νέο κανονισμό για την ε, Ευρωπαϊκή Σύνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και έκτη προτεραιότητα για τη διαδικασία στα σύνορα. Κατόπιν όριμου σκέψης προτείναμε διαγραφή και του σχετικού άρθρου για τι διατυπώσει στα σύνορα. Κρίνοντας ότι η απόφαση στην οδηγία για τις διαδικασίες που θα γίνει κανονισμός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αν ναι, τι άλλο. Οπότε πρέπει να περιμένουμε πρώτα την οριστικοποίηση του κανονισμού πριν προχωρήσουμε εμείς στον τομέα αυτό. Οι δεμοί ίσως δημιουργηθούν αντιφάσει μεταξύ των δύο λύσεων. Αυτές είναι οι έξι προτεραιότητες της ομάδας μου. Ευχαριστώ. Η Σοφή Ιντφελτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας επενέσω για το έργο σας, ε, γιατί είναι πολύ αξιόλογο και μεστό και θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις πριν σας παρουσιάσω τις ε, προτεραιότητες της ομάδας. Ξέρω ότι το τρένο έχει φύγει από το σταθμό, αλλά θα ήθελα να σημειώσω για τα πρακτικά ότι με ενοχλεί ότι έχουμε ένα πακέτο, μια δέσμη 7 προτάσεων για την εσωτερική διάσταση Τη μεταναστευτική πολιτική που έχει κολλήσει στο Συμβούλιο γιατί τα κράτη-μέλη φέρονται τελείω ανεύθυνα. Αυτό που θέλουν είναι η Ευρώπη, την Ευρώπη φρούριο. Θέλουν μια Ευρώπη φρούριο που είναι ουσιαστικά η ευρωπαϊκή εκδοχή του τείχου που θέλει να κατασκευάσει ο Τραμπ. Διαφορά δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αναδιατυπώσουμε αυτή την οδηγία. αν το αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε διαρωτώ με. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεριφέρεται ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντίθετα λαμβάνει διαταγές από τα κράτη-μέλη, κάτι που παραβιάζει τη συνθήκη. Επίσης, υπάρχει το πρόβλημα που επισήμανε η Σιλβί Ιόμ. Έχουμε επικάλυψη με άλλα θέματα που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί για κανονισμούς που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Οπότε, επίσης, έχουμε ε, συζήτηση εδώ για κάποια θέματα που ήδη έχουμε ψηφίσει και που έχουν ήδη ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο και τώρα ξεκινάμε από την αρχή πάλι για την κατάρτιση, για τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, τον κίνδυνο διαφυγής. Γιατί θα πρέπει να ε, επιληφθούμε εκ νέου για τα θέματα αυτά που ήδη έχουμε ψηφίσει. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φταίει που δεν το αποσαφήνισε στα κράτη-μέλη. Επίσης, για τι προτεραιότητε με τυχαία σειρά καταθέσαμε τροπολογίες ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις οικειοθελείς επιστροφές και λιγότερο στις κρατήσεις ή στις υποχρεωτικές ή αναγκαστικές επιστροφές γιατί τα κράτη-μέλη προτιμούν τις κρατήσεις. Αν μπορούσαν θα κρατούσαν τους πάντες. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε βιώσιμες επιστροφές, δηλαδή μεγαλύτερη υποστήριξη και μέτρα για κοινωνική ένταξη μετά την επιστροφή. Επίσης, προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών. Συμφωνώ απόλυτα ε, με τα σχόλια της ε, Μαρίας. Και να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό, γιατί αν από τη μία ε, διευκολύνουμε την κράτηση, αλλά δεν μπορούμε να κρατούμε ανθρώπους που έχουν παιδιά, τότε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να μας εξηγήσουν πώς θα βρουν την ισορροπία και πώς θα το καταφέρουν. Επίσης, προσοχή στα δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων, ΛΟΑΔΜΑ, ε, γυναίκες μόνες τους, θρησκευτικές μειονότητες, άπιστους ή άθρησκους. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της διαφυγής, θέλουμε κλειστό κατάλογο, εξαντλητικό, με ρεαλιστικά κριτήρια. Αυτό το είπαμε και στις, στην οδηγία για τις προϋποθέσεις ε, υποδοχής. Δεν θέλουμε να αφήσουμε στα κράτη-μέλη τη διακριτική ευχέρεια να ορίσουν τον κίνδυνο διαφυγής. Γιατί τα κράτη-μέλη θα κρίνουν ότι όλοι ε, ε, δημιουργούν κίνδυνο διαφυγής. Επίσης προτιμούμε ένα άρθρο για τη συνεργασία και την ενημέρωση καλύτερα, με δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά τις κοιοθελείς αναχωρήσεις, 30 ημέρες για τις οικειοθελείς αναχωρήσεις προτείνουμε με κάποιες εξαιρέσεις και σε ό,τι αφορά τα ένδικα μέσα, τις προσφυγές, προτείνουμε οι προσφυγές να διακόπτουν τη διαδικασία. Επίσης, κράτηση για λόγους δημόσιας εθνικής ασφάλειας. Απαράδεκτο. Νομίζω τα κράτη-μέλη προσπαθούν να το ε, ενσωματώσουν. Άλλωστε, εθνική ασφάλεια δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καν νομικός ορισμός τι εστί εθνική ασφάλεια. Μπορεί κάποια κράτη-μέλη να έχουν εθνικούς ορισμούς νομικούς για την εθνική τους ασφάλεια, αλλά πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε μία έννοια που είναι νομικώς απροσδιόριστη και επίσης δεν αποτελεί κοινοτική αρμοδιότητα, δεν είναι ρητή ενωσιακή αρμοδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλούμε για πολιτικέ ασύλου και όχι για εθνική δημόσια ασφάλεια. Έχουμε άλλε νομοθεσίε για τα θέματα αυτά και αν κάποιο δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια μπορεί να συλληφθεί, αλλά θα πρέπει να γίνει με διαφορετικού, για διαφορετικούς νομικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στα σύνορα και εμεί προτείνουμε διαγραφή εν ώψη της έκβασης των διαπραγματεύσεων για το σχετικό κανονισμό. Ευχαριστώ κύριε Σπινέλη. Σας ευχαριστώ, Τζούντι, εισηγήτρια. Συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση του σχεδίου εκθέσεώς σου. όσο αφορά την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη βλέπω με αρνητικό μάτι γενικά. Για λόγους παρομοίου με αυτούς που εξέφρασε η Σοφή. Δεν χρειάζεται να του απαριθμίσω, να επαναλάβω τα επιχειρήματα. Είναι τα ίδια. Ταυτόχρονα πρότεινα αρκετές τροπολογίες. Στόχος μου η ενίσχυση των εναλλακτικών που εκφράζονται από την εισηγήτρια του σχέδιου κειμένου και να στηρίξω και τις που έχουμε για να στηρίξουμε ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και συντονισμό μας με τις διεθνείς κανόνες για τα δικαιώματα των προσφύγων. Είχαμε και πληροφορίες που λάβαμε από τους εμπειρογνώμονες στα, στις πρώτες συνεδριάσεις των σκιωδών και πρότεινα γι' αυτό τη διαγραφή του άρθρου 6 όσον αφορά τον κίνδυνο διαφυγής και τη διασύνδεση που γίνεται με τη συνεργασία. Εξήγησα το σημείο αυτό. Το άρθρο αυτό πρέπει να αλλάχθει και ριζικά πρέπει να αναδιατυπωθεί. Ο ανοιχτός κατάλογος κριτηρίων όσον αφορά τον κίνδυνο διαφυγής περιέχει ε, πολλούς κινδύνους. Κίνδυνο να καλύπτονται σχεδόν όσο οι, όσοι διαμένουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας τόσο μακροσκελής κατάλογος για τον κίνδυνο διαφυγής μπορεί να έχει στα συνέπεια η απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη να είναι αυτή που συστηματικά δεν δίνει μια περίοδο για οικειοθελή αναχώρηση. Και θα κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Και τελικά θα αποφασίζεται και απαγόρευση εισόδου. Και αυτό μπορεί να αποβεί και εις βάρος τους υπηκούς τρίτων χωρών που δεν έχουν επαρκείς πόρους όσον αφορά την οικειοθελή αναχώρηση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δίνουν μια περίοδο μέχρι έξι μήνες για οικειοθελή αναχώρηση. Όσον αφορά την κράτηση στις τροπολογίες μου, ζητώ από τα κράτη-μέλη ποτέ να μην εφαρμόζουν καταναγκαστικά μέτρα, αναγκαστικά μέτρα. Και αν κάποιο κράτος μέλος απαγορεύσει να εφαρμόσει σαν τελευταίο μέσο την κράτηση, η κράτηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ειδικού ανοιχτούς χώρους και για βραχύτερες περιόδους από αυτές που αναφέρονται στην πρόταση. Αυτές οι ειδικέ εγκαταστάσεις θα πρέπει να επιτρέπουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαθήσης, να γίνονται σεβαστέα τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπηκότητων χωρών που κρατούνται και θα πρέπει το προσωπικό να είναι κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατά την άποψή μου, ποτέ δεν θα πρέπει να κρατούνται σε εγκαταστάσεις παρόμοιες με φυλακές ή σε φυλακές, αναμειγνύοντας, όπως είπε Τζούθιτ, ανθρώπους με ποινικό μητρό, με απλούς ε, παράτυπους μετανάστες που πρέπει να επιστραφούν. Για να αναδιατυπωθεί οδηγία επιστροφών και να ευθυγραμμιστεί με το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων, πρότεινα τη διαγραφή της απαγόρευσης εισόδου, άρθρο 13, διότι πιστεύω ότι η επιβολή απαγόρευσης εισόδου σε υπηκός των χωρών είναι κάτι αντιπαραγωγικό και είναι κάτι ασύμβατο με το στόχο που είναι να εφαρμόζονται οι κανόνες επιστροφής και η πολιτική επιστροφών με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και προσέθεσα σχετικές τροπολογίες, να τις συνοψίσω, η απαγόρευση κράτησης ανηλίκων και οικογενειών εν ονόματι των ε, προσόφελος των συμφερόντων του παιδιού ένα άρθρο σύμφωνα το οποίο οι των χωρών έχουν το δικαίωμα να εισακουστούν από τις αρμόδιες αρχές πριν ληφθεί κάποια ατομική απόφαση για συγκεκριμένο άτομο, δυνατότητα νομικής αρρωγής και εκπροσώπησης και γλωσσικής αρρωγής δωρεάν, εύλογο χρονικό όριο για υποβολή έφεσης κατά απόφασης επιστροφής για να εξασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος για, ε, για αποτελεσματική χρήση ενδίκων μέσων. Σύμφωνα και με αυτά που λέει η συγγήτρια, πρότεινα και εγώ μία έφεση κατά της απόφασης επιστροφής να οδηγεί σε αυτόματη αναστολή της απόφασης και σε περιπτώσεις που υπάρχουν εκρεμούσες υποθέσεις προ δικαστηρίου ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ε, η, δυνατότητα προσφυγής ε, ε, των υπόπτων και των θυμάτων ε, στα ένδικα μέσα. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος ομιλητών το Κοινοβούλιο, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το λόγο, δεν θα σας δώσω το λόγο να εξηγήσω γιατί. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να προβληματιστεί το Κοινοβούλιο περί του τι θέλει να κάνει. Είχαμε δύο συνεδριάσεις σκιωδών που καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιγράψει και να εξετάσει τη διαδικασία άρθρων προς άρθρων και είχαμε διάφορες συνεδριάσεις ήδη εδώ και συναντήσεις όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να εξηγήσει πώς ήθελε να διατυπώσει την νομοθεσία. Πιστεύω ότι τώρα δεν είναι η στιγμή για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η στιγμή για διάλογο μεταξύ ευρωβουλευτών. Και από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο θα έχει διαπραγματευτική εντολή, τότε είναι η στιγμή να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ω πρόεδρο εκφράζομαι έτσι και ωφελούμε από αυτό αυτή τη στιγμή, από τη θέση μου ως Προέδρου. Έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα. Ως εισηγήτρια να πω ότι εκτιμώ, κύριε Κοέλιο, το ότι τονίσατε τα δικαιώματα των παιδιών, όπως και άλλοι συνάδελφοι, μπορούμε σίγουρα να ενισχύσουμε τη διατύπωση της οδηγίας σχετικά. Συμφωνώ με την κυρία Ιντφέλτ ότι οι βιώσιμες επιστροφές είναι ο στόχο μας. Δεν εξετάζουμε τον αριθμό των ανθρώπων που αποχωρούν από την Ένωση. Θέλουμε αυτοί που αποχωρούν και επιστρέφουν να μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή και να μην δοκιμάσουν ξανά όταν δεν προσπαθούν να ξεφύγουν ως πολιτικοί πρόσφυγες. Συμφωνώ με την επιθυμία σας κυρία Σπινέλη πρέπει ε, να δίνονται σαφείς νομικές συμβούλες και θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω ότι θα διατυπώσουμε το κείμενο της νομοθεσίας με τέτοιο τρόπο ώστε η κράτηση που δεν μπορεί να αποκλειστεί θα είναι το τελευταίο μέσο που χρησιμοποιείται. Το έσχατο μέσο και απηχώ και εγώ τα σχόλια της κυρίας Ιντφελτ. Αυτά που είπε στην αρχή, ότι είναι αμφισβη... Δεν ξέρω γιατί κάνουμε διατύπωση οδηγίες επιστροφών. Εγώ προσωπικά να πω γιατί το κάνω. Τώρα που γίνεται είναι η δυνατότητα που έχουμε να βελτιώσουμε την οδηγία και να αλλάξουμε την εστίαση. Και δεύτερον, ακόμα δεν έχει έχει βγει εντολή από το Συμβούλιο και αυτό δείχνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο προσπαθώντας να συνεννοηθεί μαζί μας σε διάφορα θέματα ασύλου ή να συνεννοηθούν και μεταξύ για θέματα ασύλου ε, και μετανάστευση. Σε 7 Μαρτίου θα ξανασυναντηθούμε και πριν από αυτό θα σα υποβάλω συμβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώσαμε και την απογευματινή μα συνεδρίαση. Θα συναντηθούμε ξανά αύριο σε 9 η ώρα το πρωί. Γεια σα. Καλό βράδυ.